συνάδελφοι. Welcome to Libre Meeting. Καλώς ήρθατε στη συνεδρίαση της 1ης ε, Απριλίου της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Ξέρουμε ότι σε πολλές χώρες λέμε πρωταπηλιάτικα αστεία αυτή την ημέρα, αλλά η σημερινή μας συνεδρίαση είναι πολύ σοβαρή, καθόλου αστεία και ελπίζω να παραμείνετε και να ακούσετε πρώτα απ' όλα. Θα ήθελα να σας ε, θέσω υπόψη με ορισμένε αλλαγέ στην ημερήσια διάταξη. Υπάρχει το νέο σημείο 5α, ψηφοφορία από το σημείο 2 ε, Παύλα 1 του σημειώματος των συντονιστών της συνεδρίας 21η Μαρτίου σύμφωνα με τον κανόνα 205 των κανόνων του Κοινοβουλίου για το σχέδιο συμφωνίας Δανία Eurojust. Σήμερα στι 5 και 4, αν δεν ε, γίνει δεκτή η απόφαση αυτή των συντονιστών, θα μπορούσε αύριο στι 3 να λάβει χώρα η παρουσίαση του σχέδιου συμφωνίας Eurojust Δανία. Δεύτερο θέμα, το σημείο 6, ψηφοφορία επί ε, προσωρινή συμφωνία μετά από τι διοργανικέ διαπραγματεύσει για την Ευρωπαϊκή Συνορική και Εκτοφυλακή θα λάβει η χώρα αύριο στις 3 παρατέταρτο και τέλο σημείο 14 ψηφοφορία επιβεβαιωτική διεκθέσεως ε, για την πρόληψη της διάδοσης ε, τρομοκρατικού ε, περιεχομένου στο διαδίκτυο αναβάλλεται για τις 8 Απριλίου. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις προς την ημερήσια διάταξη, εγκρίνεται. Just Okay. Um, we also have some... Επίσης, έχουμε να εγκρίνουμε για κάποια πρακτικά. Από τον Ιούνιο του 18, τον Σεπτέμβριο του 18, τον Οκτώβριο του 18, τον Ιανουάριο του 19 και το Φεβρουάριο του 19. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις για τα πρακτικά θα τα εγκρίνουμε και αυτά. Επίσης, ό,τι αφορά τη διερμηνία. Για σήμερα έχουμε διαθέσιμη διερμηνία σε όλες τις γλώσσες εκτός από τα δανικά, τα κροατικά, τα μαλτέσκα και τα ιρλανδικά. Πρέπει τώρα να εγκρίνουμε τις συστάσεις των συντονιστών. και το σημείωμα τη συνεδρίας της 25 Μαρτίου για το οποίο σας μίλησα ήδη πριν. Σε αυτό το feedback note ε, λέγονται αυτά τα οποία θα πρέπει να δεχθούμε πλην του σημείου 2.1 που δυνάμει του κανόνα 205 θα συζητηθεί μας 5 και 4. Η Επιτροπή μας συμφωνεί με τις συστάσεις των συντονιστών. Ναι, από ό,τι φαίνεται. Μπορούμε λοιπόν να συνεχίσουμε εκτό από αυτό το σημείο που σα είπα. Έπειτα έχουμε να μιλήσουμε για τι κάτι εξουσιοδότηση και εκτελεστικέ πράξει. 25 Μαρτίου 2019 το Κοινοβούλιο έλαβε ένα σχέδιο εκτελεστική απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χρηματοδότηση των δράσεων τη Ένωση στο πλαίσιο του Ταμείου Ιστορική Ασφάλεια, σύνορα, θεωρήσει διαβατηρίων, έγκριση του πρόγραμματο εργασία του 2019. Η βασική νομική πράξη είναι ο κανονισμό 515-2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέση στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερική Ασφάλεια ε, του Μέσου Χρηματοδοτική Υποστήριξη ε, για τα εξωτερικά σύνορα και τι θεωρήσει, που ακυρώνει την απόφαση 574-207 EC. Η συνάδελφοι από την ΛΥΜΠΕ έλαβαν τα σχετικά μέσω του ενημερωτικού δελτίου της ΛΥΜΠΕ της 29ης Μαρτίου και υπάρχει εσωτερική προθεσμία για την κατάθεση ενστάσεως. Σε λοιπόν που κάποιος θα ήθελε να καταθέσει ε, κάποια ένσταση θα πρέπει να ενημερώσει τη γραμματεία της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ πριν τις 8 Απριλίου στις 12 το μεσημέρι. Επίσης, 25 Μαρτίου 2019, το Κοινοβούλιο έλαβε μια εκτελεστική απόφαση της Κομισιόν για τη χρηματοδότηση των δράσεων της Ένωσης στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και για την έγκριση του προγράμματος εργασίας 2019. Βασική εδώ νομική πράξη ο κανονισμός 516 2014 Έγινε λοιπόν, λάβαμε αυτή την εκτελεστική πράξη και ενημερώθηκαν σχετικά μέσω του ενημερωτικού δελτίου όλα τα μέλη της Επιτροπής μας 29 Μαρτίου. Υπάρχει εσωτερική διορία για την υποβολή ενστάσεων. Και αν επιθυμεί κάποιο να καταθέσει τέτοια ένσταση, θα πρέπει το πράξη, ενημερώνοντα τη γραμματεία πριν τι 8 Απριλίου 12 το μεσημέρι. 5 και 4 έχουμε την ηλεκτρονική ψηφοφορία και αύριο στι 3 παρατέταρτο ελπίζοντα να έχετε όλοι τις ηλεκτρονικές σας κάρτες. Και τώρα προχωρούμε με το πρώτο ουσιαστικό σημείο τη σημερινή διάταξη, που είναι το δίκτυο των ε, υπηρεσιών ε, Δικαιοσύνης και εσωτερικών Υποθέσεων θα ακούσουμε την κυρία Βιρτζίνια Λάγκμπακ, Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Σότα των Φίλων και την κυρία Κάθριν Ντεμπόλ, εκτελεστική Διευθύντρια της Europol. Σας καλωσορίζω και τις δύο Γνωρίζετε ότι εννέα υπηρεσίε Ευρωπαϊκή Ένωση που εργάζονται στον τομέα δικαιοσύνη και εσωτερικών υποθέσεων έχουν δυσπίσει ένα δίκτυο για τη βελτίωση τη διμερού και πολυμερού συνεργασία στου τομεί κοινού ενδιαφέροντο. Η αιτήσια έκθεση ε, του 2018 σε σχέση με ε, τα πεπραγμένα του δικτύου δημοσιοποιήθηκε το Φεβρουάριο και περιλαμβάνεται στο φάκελο των εγγράφων της συνεδρίασης. Κυρία Λάγκμπακ θα μας παρουσιάσει λοιπόν ε, την επισκόπηση των βασικών επιτεγμάτων της περσινής χρονιάς και εν συνεχεία θα δώσω το λόγο στην κυρία Ντεμπόλ που είναι η διευθύντρια του δικτύου για να μας παρουσιάσει τις προτεραιότητες του 2019. Και επειδή είμαι εδώ κυρία Λάγκμπακ σήμερα, καλέσαμε και τα μέλη της Επιτροπής Γυναικών Κύριε Λάγκμπακ, έχετε το λόγο. Ζητώ συγγνώμη που δεν είναι γεμάτη αίθουσα, απλά πολύ συνάδελφοι ακόμη είναι καθοδόν. Έχετε το λόγο λοιπόν. Καλησπέρα σας μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ και της Επιτροπής ΦΑΜ. Το πρωί σκεφτόμουν ότι για μένα είναι μια σπάνια δυνατότητα. Γυναίκες και διευθύντριες σε οργανισμούς για την ε, δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις να είμαστε εδώ ταυτόχρονα σήμερα. Και δεν είναι και φάρσα, τα πράγματα αλλάζουν. Την τελευταία φορά που συζητήσαμε πριν από ένα χρόνο περίπου είχα υποσχεθεί ότι κάτι θα αλλάξει σε σχέση με, τις, με τον Οργανισμό της Δικαιοσύνη και των Ιστορικών Υποθέσεων, λόγω της εντολή μας και των προσπαθειών που έχουμε καταλάβει, καταβάλει, συγγνώμη, να προσθέσουμε και ένα ανθρώπινο πρόσωπο, την ανθρώπινη διάσταση στις κλίμακες των υπολογιστών, τι κολόνες και τι στατιστικές που είναι τόσο τεχνικά. Ε, νομίζω ότι κάτι καταφέραμε και μάλιστα καλά. Το Παράρτημα 3 σας λέει περισσότερα για τις λεπτομέρειες το τι γίνεται με τις γυναίκες, άντρες, κορίτσια και αγόρια που είναι η ουσία της έκθεσης. Τώρα όμως αν ναι, έχετε για να το καταλάβετε καλύτερα και να μπορείτε να το διαβάσετε, έχουμε το παράρτημα 1 όπου απαριθμώνται όλες μας οι δραστηριότητες και περιγράφονται κατά Αλλά για να ανακεφαλαιώσω, το σύνολο των δραστηριοτήτων του οργανισμού, για να μπορείτε να τα διαβάσετε μετά μόνοι σας κατά θα πω το εξή, από την επόμενη διαφάνεια. Από πέρσι έχουν συμβεί τα εξή. Έχουμε το θέμα, τις θεματικές και ειδική στόχευση, καθώς και οριζόντια δουλειά. Για να ενισχύσουμε την τεχνική διάσταση και τις δραστηριότητές μας, συνεργαζόμαστε ε, με όποιον είναι αρμόδιος βάσει της εντολής μας και προσπαθούμε να προσθέσουμε και ειδικά στοιχεία λόγω χάρη για το πώς η ασφάλεια και η μετανάστευση πρέπει να αντιμετωπιστούν, τι προκλήσεις μπορεί να προκύψουν ή ξέρω εγώ για την στρατηγική της μετανάστευσης και της ασφάλειας τι πρέπει να κάνουμε. Δείτε τα και στην έκθεση. Από τη δική μας την πλευρά προσπαθούμε να δώσουμε έμφαση στο που γίνεται να προβάλλουμε τη δουλειά των ανδρών και γυναικών στην ασφάλεια, τη ριζοσπαστικοποίηση, την εμπορία. Όλοι επηρεάζονται με διαφορετικό τρόπο και άντρε και γυναίκε, κορίτσια και αγόρια. Έχουμε ξεκινήσει λοιπόν κατά αυτόν τον τρόπο και θα ε, εντείνουμε τι προσπάθειέ μα, διότι είναι η πρώτη μα προσπάθεια. Αν κανεί δεν προσπαθήσει, δεν μπορεί και να δει τι δεν πετυχαίνει. Η ανταλλαγή πληροφοριών και η ενημέρωση ήταν ένα άλλο τομέα όπου είδαμε ότι εάν δράσει κανείς εγκαίρος, εντοπίζει κάποιες αρνητικές τάσεις και μπορεί να τις αναχαιτήσει. Επίσης, αν συνεργαστεί με άλλους φορείς εγκαίρος, οι αποφάσει λαμβάνονται πιο τεκμηριωμένα, πιο υπεύθυνα και έχουν καλύτερο αποτέλεσμα. Ανταλλαγή λοιπόν πληροφοριών. Σημαντικό κομμάτι του έργου μα. Συζητήσαμε και με τρίτε χώρε. Και ω προ τα δικά μα, γιατί αυτά γνωρίζω καλύτερα, ω προ τον ακροτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων, Εάν ε, πάρει κανεί τις γνώσεις και τι εμπειρίε των συνοριοφυλάκων ή άλλων ελεγκτών ή όσων ασχολούνται με την ένταξη στα μεταναστευτικά κέντρα, μπορεί να καταφέρει να συγκεντρώσει στοιχεία και να αλλάξει τη ζωή κάποιας κοπέλας που θα μπορούσε να υποστεί ε, κλειτοριδεκτομή. Για την στοχευμένη εκπαίδευση. Αυτό το αναλαμβάνει συνήθω ο ΣΕΠΟΛ, αλλά σε συνεργασία και με πολλούς άλλους οργανισμούς ώστε να αντιμετωπιστούν οι ειδικέ ανάγκες που έχουν ε, ήδη οριστεί από την αρχή. Ως προς την ισότητα των φύλων. Τι κάναμε. Όπως έχουμε πει, νομίζω πολύ είναι επιφυλακτική ή διστακτική όταν μιλάμε για τον ευθυγραμμισμό της διάστασης των φύλων. Αλλά εάν δεν το κάνει κανείς δεν ξέρει και τι χάνει. κάτι που ξεκινήσαμε και έτυχε πολύ καλή υποδοχή από τους υπόλοιπου οργανισμούς ήταν ότι εάν δεν γνωρίζει κανεί τα κοινά και τι ελλείψει, εάν δεν γνωρίζει τι τάσει υπάρχουν στο ευαίσθητο θέμα των φύλων, οι στατιστικέ δεν ορίζονται με βάση το φύλλο, δεν συγκεντρώνουν στοιχεία με βάση το φύλλο. Οπότε δεν ξέρει κανεί ε, τι συμβαίνει, ποιο πλήττεται περισσότερο, ποιε είναι οι τάσει. Αποφασίσαμε λοιπόν με ένα εργαστήριο για, όλες, για όλου του οργανισμού ταυτόχρονα να δούμε τι γίνεται με του ανθρώπου που παίρνουν μέρο σε επιχειρήσει. Είδαμε τι διαφορά υπάρχει, ε, ποια είναι τα στοιχεία Ε, τι στατιστικά δεδομένα υπάρχουν και έτσι οργανώσαμε τις συζητήσει μας. Περισσότερο οι περισσότεροι από τους οργανισμούς μας, όσοι συμμετέχουν στο δίκτυο, βλέπουν την αξία της δράσης μας, διότι η δική μας δουλειά είναι να αναφέρουμε τι συνέβη σε εσά, πώς προχωρήσαμε, πώς ε, λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι πρέπει να χρηματοδοτεί, πώς επηρεάζει τη ζωή αγοριών και κοριτσιών στην πράξη. Πρέπει να ξέρουμε πόσα αγόρια και πόσα κορίτσια όμως επηρεάζονται. Αυτό είναι μέρος της δουλειά μας και θα συνεχίσουμε Χωρί σταματημό. Γιατί είναι σημαντική η βάση δεδομένων που θα δημιουργήσουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση για τα δεδομένα τη ευθυγράμμιση του φύλου, τη διάσταση του φύλου. Θα μπορούσαμε λοιπόν ε, με κοινέ προσπάθειε να φέρουμε πραγματική αλλαγή. Η έκθεση ω προ το παράρτημα 3 που το συμφωνήσαμε αφού το συζητήσαμε με όλου του οργανισμού ήταν για να φωτίσουμε ένα συγκεκριμένο τομέα και επιλέξαμε τον τομέα που είναι το μέλλον που μπορεί να παρουσιάσει όχι μόνο κινδύνου, αλλά και μεγάλο δυναμικό και δυνατότητε ανάπτυξη δουλειά και έκφραση στον πολιτικό βίο, έκφραση την κοινοβουλευτική σας δουλειά και στην ψηφιοποίηση. Αυτό που ε, αναλύσαμε λοιπόν, ότι κοιτάξαμε πώς η ψηφιοποίηση, η ψηφιακή δηλαδή διάσταση, επηρεάζει ξεχωριστά γυναίκες και άντρες. Ποιες είναι οι διαφορές, ποιες είναι οι δυνατότητες κοιτάξαμε τι μπορούμε να εντοπίσουμε και να στοχεύσουμε με ευρωπαϊκά κονδύλια ώστε να αναπτυχθεί περαιτέρω. Ε, τι θα θέλαμε να γίνει ιδανικά μας ε, απασχόλησε. Επίσης στην έκθεση αν τη διαβάσετε θα δείτε και άλλες διαφορετικές διαστάσεις όπως την εμπορία ή το κυβερνό έγκλημα ή την συμμετοχή στον πολιτικό βίο. Ας πούμε, στην έκθεση φαίνονται διαφορετικές διαστάσεις ε, που μπορούν ε, να αναλάβουν δράση διάφοροι οργανισμοί για τα αγόρια και τα κορίτσια. Υπάρχει διαφορά προς το φύλλο, υπάρχει διαφορά και στην ψηφιοποίηση. Είναι μεγάλες οι αποστάσεις αυτή τη στιγμή και για την ώρα ε, οι γυναίκες χάνουν. Οπότε στην έκθεση μπορείτε να δείτε περισσότερα. Προτείνουμε πολλά πώς ε, τα θεσμικά όργανα, οι εθνικοί φορείς, τα ευρωπαϊκά όργανα μπορούν να ανταποκριθούν με διαφορετικούς τρόπους. Προκειμένου η δουλειά αυτή να γίνει πραγματικά επικοδομητική για όλους, και άνδρες και γυναίκες, αγόρια και κορίτσια. Και όπω έχετε πει, έχει, όπως έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν, πολλή κουβέντα έχει γίνει για τη σεξουαλική παρενόχληση. Οπότε αυτό αποσχολεί όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά οργανά και του φορεί, αλλά περισσότερο ασχολούμαστε με του οργανισμού δικαιοσύνη και ιστορικών υποθέσεων. Κοιτάζουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε το θέμα σωστά, εγκαίρω και με πρόληψη. Αυτό είναι ο γνωμονά μα. Ε, μηδενική ανοχή κάναμε μια τέτοια δήλωση μηδενική ανοχή που λέγεται ότι όλοι οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί και ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα υπογράφουν. Συζητήσαμε με όλου του διευθυντέ και είχαμε και ένα σεμινάριο εμπιστευτικό και απόρριτο όλων των συνεργατών ε, και συμβούλων που ασχολούνται με το θέμα αυτό και το Κοινοβούλιο έχει τέτοιον. Είναι πολύ ενδιαφέρον να δει κανεί πώ βλέπει κανείς να εξελίσσει τη δουλειά αυτών των συμβούλων όταν αρχίσει να το προωθεί το θέμα από πάνω προς τα κάτω. Δεν πάει χαμένη η δουλειά τους και εμείς τους υποστηρίξαμε. Έχουμε επίσης και το εργαστήριο για το μέσο management και τους ανθρώπινους πόρους. Κοιτάξαμε να ετοιμάσουμε υλικό που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τουλάχιστον οργανισμοί και ελπίζω και το Κοινοβούλιο. το ίδιο πλαίσιο σας αφορά και εσάς. Μπορείτε να αλλάξετε διαφάνεια παρακαλώ. Και τώρα τα διδάγματα που αντλήσαμε. Ένα από τα βασικά μας ευρήματα κατά τη συνάντηση των διευθυντών τον Νοέμβριο ήταν ότι ήταν ότι όλοι γνωρίζουν και η Επιτροπή Λίμπα ακόμη περισσότερο ότι το τι κομμάτι του προπολογισμού και ετησίω και στο επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο αναλογή στα θέματα αυτά, δικαιοσύνη, στου οργανισμού δηλαδή δικαιοσύνη και εσωτερικών υποθέσεων, είναι σημαντικό. Δυστυχώ δεν έχουν ωφεληθεί αρκετά όλοι οι οργανισμοί. Κάποιοι έχουν νέε αρμοδιότητε. Χρειάζονται νέα στήριξη από τον προπολογισμό. Κάτι που είναι φυσικό και εύλογο. Όμω, άλλοι έχουν μεγαλύτερε ανάγκε και περισσότερε αρμοδιότητε. Σε κάποιου οργανισμού ανατίθενται περισσότερα, απαιτούνται περισσότερα, αλλά δεν υπάρχει απαραίτητη πρικοδότηση. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη δυσκολία. Πώ μπορούμε να υποστηριχθούμε εδώ, τεχνολογικέ εξελίξει. Εδώ η έκθεση εντοπίζει ότι υπάρχουν νέα στοιχεία, νέα ε, σύνορα τεχνολογικών εργαλείων που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν καλύτερα για όλου του οργανισμού αυτό μπορεί να είναι και πλεονέκτημα αλλά και πρόβλημα. Για τι τρίτε χώρε. Συζητήσαμε πώ μπορούν οι οργανισμοί να συνεργαστούν καλύτερα. Έχουμε τη δική μα εντολή και ε, συνεργαζόμαστε κάποιε φορέ παράλληλα με κάποιου οργανισμού τρίτων χωρών. Όταν ανταλλάσσουμε πληροφορίε το βλέπουμε αυτό. Θα μπορούσαμε ενδεχομένω να αναπτύξουμε για κοινά προγράμματα γιατί κάποιε φορέ Θέλει κανείς αυτό το επιπλέον, να κερδίσει ένα χαμόγελο, να κάνει κάτι το καινούργιο έστω και αν είναι μικρό και για την προστιθέμενη αξία. Έχουμε συνεργαστεί με το δίκτυο των οργανισμών για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά βάσει τη εντολή μα. Με τελείω διαφορετικέ ιδέε και πράγματα. Όμω πρέπει να δείξουμε και στου Ευρωπαίου πολίτε, όχι μόνο στο Ευρωκοινοβούλιο, στου ανθρώπου, στου καθημερινού, ποια είναι η προστιθέμενη αξία τη δουλειά μα. Αυτά λίγο πολύ είναι όσα έχουμε. Τελευταία διαφάνεια. Τι πετύχαμε την τελευταία χρονιά. Θα συνεχίσουμε βεβαίως, αλλά από τη δική μου την πλευρά χαίρομαι πάρα πολύ που επιτέλους ξεκινήσαμε να σκεφτόμαστε το θέμα άντρες και γυναίκες, αγόρια και κορίτσια και ξέρουμε ότι είναι πολύ διαφορετική. Εάν αγνοούμε τις διαφορές ποτέ θα πετύχουμε όσα επιθυμούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την επισκόπηση, την εξαντλητική. Ήδη ε, έχω σκεφτεί κάποιες ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση αυτή. Θα δώσω μέσα στο λόγο στην κυρία Ντεμπόλ για 10 λεπτά περίπου. Ευχαριστώ. Thank you and thank you for giving me the opportunity to... Ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να σας ενημερώσουμε για τις προτεραιότητες που έχουμε ε, ε, ως Προεδρείο των ε, οργανισμών αυτών για το 2019 που έχουν σχέση με τη δικαιοσύνη και τα εσωτερικά και η ποικιλομορφία και η συμπερίληψη και η άρση των αποκλεισμών για μας πολύ σημαντική. Και χαίρομαι που καλωσορίζουμε σήμερα εδώ όχι μόνο τα μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ αλλά και της Επιτροπής ΦΑΜ. Βασική προτεραιότητα στην οποία συμφωνήσαμε στους οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα εσωτερικών και δικαιοσύνης είναι ότι θέλουμε να προβληματιστούμε σε στρατηγικό επίπεδο για το ρόλο των οργανισμών μας και τη συνεργασία μεταξύ τους. Πώς εντασσόμαστε στην ε, ε, στρατηγική και την ατζέντα της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. στο τέλος της Προεδρίας θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα. Για να ορίσουμε το πλαίσιο των συζητήσεων ε, στο δίκτυό μας, ε, αποφασίσαμε ποια είναι τα σημεία που μας ενδιαφέρουν ε, όλους. Διαλειτουργικότητα των συστημάτων πληροφόρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη συνέχεια ρόλος και θέση των οργανισμών στο τοπίο ασφάλειας Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεταξύ αυτών θέματα κοινού ενδιαφέροντος και κοινών ανησυχιών με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και το τρίτο είναι η ε, διάδραση και ενδεχομένως και συνέργειες με άλλους οργανισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός του πεδίου εσωτερικών και δικαιοσύνης. Επίσης έχουμε προσθέσει και κάποια θέματα ad hoc που είναι η χρηστή διακυβέρνηση ε, στον τομέα και στους οργανισμούς μας και μπορούμε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν πώς μπορούν οι οργανισμοί μας να αντιμετωπίσουν το θέμα της καινοτομίας, γιατί η Europol, Φερρυπίν, είναι ε, βασικός στρατηγικός στόχος μας αυτός για το μέλλον, καινοτομία. Η δική μας υπηρεσία, ο οργανισμός μας, σε συνεργασία με τους άλλους, θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε να καινοτομούμε από κοινού. Τρίτο θέμα, ευκαιρίες και προκλήσεις ε, στην ε, χρηματοδότηση ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το τελευταίο είναι η ε, διαφορετικότητα, η ε, ποικιλομορφία και η άρση των αποκλεισμών. Όλα αυτά θα τα δούμε στις... Μάλλον τα είδαμε στις 23 Νοεμβρίου του 2018 και θα τα επεξεργαστούμε και στη συνέχεια. Όπως σας είπα, έχουμε προγραμματίσει σε επίπεδο εργασίας τρεις συνεδριάσεις του δικτύου. Βλέπετε στη διαφάνεια τις ημερομηνίες. Επίσης, στις 22 Νοεμβρίου 2019 θα συναντηθούμε επικεφαλής των οργανισμών αυτών. Εκτός αυτών των συνεδριάσεων, έχουμε και συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων που διοργανώνουμε σε έξι τομείς που θα καλύψουν οι συνεδριάσεις των εμπειρογνωμόνων. Θέματα ε, τεχνολογίας προφορίας και κυβερνοασφάλειας, επικοινωνία, εξωτερικές σχέσεις ε, των οργανισμών και πώς μπορούμε καλύτερα να συνεργαζόμαστε και πιο στενά, ε, διαφορετικότητα, συμπεριλήψη, ένταξη, εκπαίδευση, πάρα πολύ σημαντικό κατάρτιση, πώς μπορούμε να τη μεταξελίξουμε και πώς μπορούμε να συνεργαζόμαστε στα θέματα αυτά ε, δικαιοσύνης και ε, εσωτερικών και προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τεράστιο ζήτημα για όλες τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς. Ε, ακόμα είναι που συζήτηση ημερομηνίε των συνεδριάσεων των εμπειρογνωμόνων. Τα αποτελέσματα αναμένονται ε, να ε, υποβληθούν στα τέλη του 19 υπό τη μορφή ενός στρατηγικού έγγραφου. Το έγγραφο αυτό θα το συνυποβάλλουμε με την ετήσια έκθεση που κάνουμε στην Επιτροπή Κόζη ε, και θα παρουσιαστεί του χρόνου στις αρχές του έτους στην Επιτροπή σας. Λίμπε για να ε, γνωρίζουν οι νομοθέτες ε, ε, ποιες είναι οι τρέχουσες στρατηγικές ανάγκες των οργανισμών αφενός και αφετέρου πώς μπορεί να ενισχυθεί περισσότερο η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων αυτών οργανισμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το στρατηγικό έγγραφο φιλοδοξεί να τροφοδοτήσει την πολιτική συζήτηση από τη σκοπιά, ε, την επιχειρησιακή όπως τη βλέπουμε εμείς στους οργανισμούς. Τα επόμενα λίγα έτσι θα είναι σημαντικά για μας έτσι ώστε να ορίσουμε το ρόλο ορισμένων οργανισμών μας και να δούμε και ποια προβλήματα υπάρχουν και προκλήσεις. Τα ε, ανέφερε και η Virginia Langback για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο που φυσικά έχει επίδραση στη λειτουργία των οργανισμών. Ε, αυτό το στρατηγικό έγγραφο πιστεύω θα βοηθήσει και το νέο κοινοβούλιο να κατανοήσει καλύτερα ε, το ρόλο και το έργο των διαφόρων οργανισμών και την καινούργια έκθεση COSI έτσι ώστε να γνωρίζουν καλύτερα ε, πώς ε, έχει καλή συνεργασία μεταξύ των οργανισμών στο δίκτυο, ενδεχομένω να προκύψουν και κάποιες συστάσεις που ε, θα θέλουν να εξετάσουν οι Επιτροπές Κόζη και η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Θέλω να σας ευχαριστήσω ως Επιτροπή Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Γιατί οι συζητήσεις που είχαμε μαζί σας, πιστεύουμε, και η διάδραση που είχαμε ε, με την Επιτροπή σας είναι πολύτιμα ε, στοιχεία για την ε, Europol. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη και στη δημοσιονομική συζήτηση. Το Κοινοβούλιο επένδυσε πολύ πολιτική ενέργεια για να προωθήσει τα θέματα των οργανισμών μας και εντός φυσικά των αρμοδιοτήτων του ε, στην υπηρεσία των Ευρωπαίων πολιτών. Επιστεύω ότι ε, αυτά ε, και χειροπιαστά αποτελέσματα έχουν ήδη προκύψει και πραγματικά είμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τη Βιρζίνια Λάγκμπακ για την περσινή προεδρία της και για την εξαιρετική εργασία της στη θέση αυτή και ως πρόεδρος του δικτύου οργανισμού με χαρά να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και την Καντεμπόλ. Βολιδοσκοπώ σκοπό για να δω ποιοι θέλουν να πάρουν το λόγο. Αλλά πριν από αυτό, για τις δύο παρουσιάσεις, ε, θέλω να πω ότι αυτό που φαίνεται είναι ότι με την ιδιότητά σας και οι δύο προσπαθείτε να ευαισθητοποιήσετε και να προωθήσετε ιδέες ε, για τη συνεργασία και τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σε θέματα ισότητα των φύλων ε, που έχουν να κάνουν με το φύλλο αλλά και σε ό,τι αφορά τη διαλειτουργικότητα, την προστασία δεδομένων και πάντοτε με γνώμονα τη βελτίωση της συνεργασίας ε, του έργου των διαφόρων οργανισμών. Ως πρώτη ερώτηση θα ήθελα να επανέλθω σε αυτή την προσέγγιση βάση φύλου και το θέμα της ψηφιοποίησης. Οι απόψεις δίστανται όταν μιλάμε για την ψηφιοποίηση. Δυστυχώς, εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές. Και θα ξεκινήσω με ένα έτσι παραδοσιακό παράδειγμα ότι τα κορίτσια πρέπει να παίζουν με κούκλες και τα αγόρια με αυτοκίνητα και ούτω καθεξής και έτσι μεγαλώνουν και συνεχίζουν οι ρόλοι να διονίζονται. Με την ψηφιοποίηση οι ιδέες αυτές μένουν, υπάρχουν στο ψηφιακό περιβάλλον ή υπάρχει κάτι διαφορετικό. Υπάρχουν διαφορετικές δηλαδή δυνατότητες για μια διαφοροποίηση στα παραδείγματα και τους ρόλους που λαμβάνουν τα δύο φύλλα. Ναι, ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Πράγματι, αυτό κάναμε ακριβώς. Αναλύσαμε τι κάνουν τα κορίτσια και τα αγόρια. Η νέα γενιά πρέπει να σας πω πως είναι η πλέον προχωρημένη σε ό,τι αφορά δηλαδή, τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων. Και δεν υπάρχει και σχεδόν καμιά διαφορά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης ε, και τα σχετικά. Όταν αρχίσουν να επιλέγουν δε το αντικείμενο των σπουδών τους, αυτά τα στερεότυπα που αναφέρατε, ότι δηλαδή το αγόρι θα πρέπει να κάνει αυτό, το κορίτσι το άλλο, ε, ήδη βλέπουμε τα πρώτα συμπτώματα ε, κοινωνική λειτουργή, κοινωνικές υπηρεσίες είναι κάτι που προτιμούν οι γυναίκες και τα αγόρια ενθαρρύνονται να σπουδάσουν ε, πολιτική μηχανική, μηχανολόγοι κτλ. 70% των ε, φοιτούντων ε, όμως σε τεχνολογικά ιδρύματα είναι αγόρια και τα υπόλοιπα είναι κορίτσια. Και το 2025 θα έχουμε 8% γυναίκες, ε, γυναικολόγους, ε, ε, συγγνώμη, μηχανολόγους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λοιπόν ήδη ένα πρόβλημα. Πρέπει να αλλάξουν τα πρότυπα και να επιλέγουν διαφορετικά οι κοπέλες γιατί αλλιώ έχουμε πρόβλημα ανταγωνιστικότητα. Ε, το ποσοστό πριν δεν ήταν 70%, ήταν 7%. Επίση, η παρενόχληση, ο κτλ. Ε, όλα αυτά έχουν ριζωμένε ε, αιτίε στην παιδεία, ίσως στο πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά. Δηλαδή έχουν ευθύνες οικογένειες, οι γονείς και τα σχολεία κοινωνία γενικότερα. Αν δούμε όμω τι γίνεται στο διαδίκτυο με τι ψυχικέ τεχνολογίε, ακόμη και κάποιο πει ότι ε, ναι μεν μπορεί να μην υπάρχουν εθνικοί φραγμοί και μπορεί κανεί να εκφραστεί ελεύθερα και μάλιστα προ όλο τον κόσμο, τα κορίτσια μετωπίζουν παρόλα αυτά πολύ περισσότερε απειλέ. Παρενοχλούνται με τον, άλλο τρόπο, ε, υπάρχει έλλειψη σεβασμού, άρα εκτίθενται πολύ περισσότερο στη βία σε σχέση με τα αγόρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Άρα έχουμε να κάνουμε ακόμη πολλή δουλειά. Παρότι 100 χρόνια τώρα έχουν δικαίωμα ψήφου γυναίκε. Δεν αρκεί αυτό όμω. Υπάρχουν ακόμη πολλέ διαφορέ μεταξύ των δύο φίλων. Κυρία Ντεμπόλ, θα θέλω να απαντήσει κάτι τώρα. Γιατί, για να μην ειλικρινή, εκπλήσωμαι και με τον εαυτό μου κάποιε φορέ. Όταν βλέπω πόσε υπηρεσίε και πόσου οργανισμού έχουμε στην Ευρώπη. Υπάρχουν κάποιοι μεγαλύτεροι που του ξέρουμε όλοι και κάποιοι μικρότεροι. Προσπαθούμε να βελτίσουμε τη συνεργασία μεταξύ των διαφορών οργανισμών. Εσείς βλέπετε κάποιες συγκεκριμένες προκλήσεις για ορισμένους οργανισμούς και ιδίως τους μικρότερους, για τους οποίους ίσως τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα από ότι για τους μεγαλύτερους ε, να αναπτύσσουν σχέσεις τα κτλ. Βλέπετε κάποιες ειδικέ προκλήσεις μήπως. Ευχαριστώ. Στους οργανισμούς δικαιοσύνης και εσωτερικών είναι πολύ σημαντικό ο καθένας να γνωρίζει ποια είναι η θέση του στο θεματολόγιο της ασφάλειας και ο ρόλος του. Έχουμε λοιπόν καλή συνεργασία πιστεύω, ειλικρινή συζήτηση για το ποια είναι τα βασικά ε, που μπορούμε από κοινού να ε, εκτελούμε, ποιοι είναι οι πόροι που έχουμε, κυρίως και οι μεγάλοι οργανισμοί, θα πρέπει να υποστηρίζουν τους μικρότερους για τη βασική δουλειά. Ας πούμε, ΣΥΠΟΛ και Europol. Ε, ΣΥΠΟΛ είναι αστυνομική ε, ε ακαδημία αλλά δεν μπορούν από μόνοι τους να επομιστούν αυτό το έργο. Ε, το πρώτο δεκάμινο όταν ανέλαβα έκανα μια περιοδία σε όλα τα κράτη-μέλη και όλες οι ε, διοκτικές αρχές ζητούν επιπλέον κατάρτιση. Έχει αναλάβει λοιπόν η Ευρωπαϊκή ε, Αστυνομική Ακαδημία, η ΣΥΠΟΛ, αλλά και ο Frontex και η Europol. Θα πρέπει να τους υποστηρίζουμε με πραγματογνώμονες, με εμπειρογνώμονες δικούς μας αλλά και των εθνικών αρχών και με τη Virginia Langback έχουμε πολύ καλή συνεργασία, διότι συνεργαζόμαστε και εμείς σε θέματα ισότητας φύλου και ισορροπίας και χρησιμοποιούμε τη δική τους πραγματογνωμοσύνη. Δεν χρειάζεται να ξανακάνουμε εμεί τι ίδιε μελέτε. Ε, πρέπει να υπάρχει αυτή η διαλειτουργικότητα και να ξέρουμε και να αναγνωρίζουμε ποιο είναι ο ειδικό σε κάθε τομέα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Σίπελ. Ε, πολύ χρήσιμο αυτό. Παρόλο που απομένει ακόμα πολλή δουλειά να γίνει. Σα ευχαριστώ για το έργο σα. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Λάγκμπακ. Καλή επιτυχία στο μέλλον, διότι τώρα Ε, είστε στη δεύτερη και τελευταία θητεία σας ε, που τελειώνει ενώ η κυρία Ντεμπόλ ε, θα ξανάρθει του χρόνου στην Επιτροπή Λίμπε να μας τα πει. Σας ευχαριστώ που ήρθατε και δυο σας και καλή δύναμη στο έργο σας ό,τι και να κάνετε. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.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 Μπορούμε να περάσουμε αμέσω στο επόμενο θέμα, στην ημερήσια διάταξή μας. A Βλέπω διάφορες συνομιλίες, αλλά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 Λοιπόν, τώρα είμαστε στην επόμενη επιτροπή, ΚΟΖΗ, μόνιμη επιτροπή επιχειρησιακής συνεργασίας σε θέματα εσωτερική ασφάλειας και θα ακούσουμε την παρουσίαση, την έκτη ε, έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια για τα πεπραγμένα της Επιτροπής αυτής για την περίοδο Ιουλίου 2017-Δεκεμβρίου 2018 από τον προσκεκλημένα μας, τον οποίο και καλωσορίζω στην Επιτροπή μας, τον κύριο Βίκτορ Βίλια Προετέζη από τη Ρουμανική Προεδρία του Συμβουλίου και πρόεδρο της Μόνιμης Επιτροπής Επιχειρησιακή συνεργασία. Καλωσορίσατε στην Επιτροπή μας, θα μας παρουσιάσετε την έκτη έκθεση η οποία δείχνει την επιχειρησιακή δραστηριότητα στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας, αλλά επίσης και την εδραίωση ε, του ρόλου της Επιτροπής Κόζη σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας. Επίσης, η έκθεση δείχνει ότι υπάρχει πρόοδος για την επίτευξη της συνέργειας μεταξύ ε, της Europol και της Κόζη για, την εκτίμηση κινδύνου και αυτό πολύ σημαντικό και γενικά πώς συνεργάζεται με τους γενικούς διευθυντές τελωνίων, με τους επικεφαλείς των διαφόρων αστυνομικών υπηρεσιών και άλλες αρμόδιες αρχές. Ε, χωρίς ε, περαιτέρω καθυστέρηση θα δώσω τώρα το λόγο για 10 λεπτά και στον κύριο ε, Απροϊτέζη. Thank you very much. Uh, is doing a lot of work, so I will try to be... Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολλά αυτά που θα είχα να πω. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται πιο σύντομος, ε, αλλά συνεκτικός. Ευχαριστώ για τη χαρά ε, που έχω και το προνόμιο να σας ενημερώνω υπό την ιδιότητά μου του Προέδρου της Επιτροπής Κόζη σχετικά με τα πεπραγμένα μας σε σχέση με την εσωτερική ασφάλεια και την επιχειρησιακή συνεργασία. Θα ήθελα να σας δώσω μια επισκόπηση για τις βασικές ε, δραστηριότητες και τα αποτελέσματα της περίοδου Ιουλίου 2019. 17 Δεκεμβρίου 2018. Κυκλοφόρησε η έκθεση και την έχετε λάβει σύμφωνα με το άρθρο 71 της συνθήκης. Το τρίο ήταν Εστονία, Βουλγαρία και Αυστρία στις Προεδρίες και η Επιτροπή Κόζη εξακολούθησε να λειτουργεί ε, για το σκοπό που είχε ιδρυθεί για την καλύτερη συνεργασία και συντονισμό της εσωτερικής ασφάλειας. Επειδή είναι πολύ ευρύ το πεδίο η Επιτροπή ΚΟΖΗ έχει ρόλο συμβουλευτικό ε, επιτήρησης και λήψης αποφάσεων ε, με ε, πυρογνώμονες από όλα τα κράτη-μέλη και όταν χρειάζεται προσκαλούνται και οι οργανισμοί που ασχολούνται με θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών και που ακούσαμε προηγουμένως. Είναι η πλατφόρμα σε πολλά θέματα και σε πολλούς οργανισμούς αστυνομία, τελωνία, συνοριοφυλακή, δικαστικές αρχές και, και εκπαίδευση αστυνομικών. Έχετε αρκετό χρόνο, δεν χρειάζεται να τα διαβάζετε με τέτοια ταχύτητα, λέει ο Πρόεδρος. Μάλιστα. Αυτή ήταν η περίοδο λοιπόν και οι δραστηριότητε. Σήμερα από την έκθεση αυτή, εγώ θα ήθελα να επικεντρωθώ σε έξι βασικού τομεί. Το κύκλο πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα, η καταπολέμηση τη διακίνηση ε, μεταναστών, ε, συμμετοχή των τελωνίων στην εσωτερική ασφάλεια, αντιμετώπιση τη τρομοκρατία, ε, ηλεκτρονικό έγκλημα και η ε, ε, σχέση εσωτερικής με εξωτερική ασφάλεια. Η ΚΟΖΗ έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίζει ε, στην πολιτική μας που λέγεται και impact για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τότε που ιδρύθηκε το 2010 δίνει το τον για να αντιμετωπίζουμε τις βασικές απειλές στην ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα και στη χρήση και στη συγκέντρωση όλων των διαφόρων ενδιαφερομένων από διάφορες υπηρεσίες και οργανισμούς και με διαφορετικά εργαλεία και δραστηριότητες για να αντιμετωπίζουμε τις προτεραιότητες μας σε σχέση με το έγκλημα. Τον Ιούνιο ε, στο Συμβούλιο Ιστορικών και Δικαιοσύνης ε, επανέλαβαν τη δέσμευσή τους οι Υπουργοί προς την κατεύθυνση αυτή. Είναι μια κοινή πλατφόρμα συνεργασίας για ένα ευρύ ε, κύκλο ενδιαφερομένων, πολυεπίπεδη απάντηση ε, σε περίπλοκες καταστάσεις σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος. Η ΚΟΖΗ λοιπόν έχει ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο πολιτικής με εξαιρετικά αποτελέσματα και αναμένεται ο επόμενος τώρα για την περίοδο 2018-2021. Για να σας δώσω μερικά παραδείγματα, οι κοινέ μέρες δράσης που είναι σαφής ε, ένδειξη της επιτυχίας μας ε, υπό τη στρατηγική ε, καθοδήγηση της ΚΟΖΗ. Από το 2017 μέχρι και το 2018 1.630 περιπτώσεις και έρευνες ξεκίνησαν, υποθέσεις στη δικαιοσύνη. 433 ε, όπλα κατασχέθηκαν και εντοπίστηκαν 1.528 θύματα διακίνησης, καθώς επίσης και συνελήφθησαν 2.270 ε, ύποπτοι. Ε, καταλαβαίνετε ότι ενισχύεται έτσι η ευρωπαϊκή πολιτική. Έχουμε και νέο ε, μηχανισμό αναφορών βελτιώνουμε την επικοινωνία στα επιχειρησιακά αποτελέσματα. Αυτό ήταν ιδιαίτερα ε, ενδιαφέρον αυτή την περίοδο. Υπάρχει και μια σειρά συστάσεων για την επικοινωνία και τη βελτίωση της προβολής ε, με ένα νέο λογότυπο. Ένα δεύτερο που θα ήθελα να σας αναφέρω και να σας ενημερώσω κατά πολέμηση της διακίνησης μεταναστών. Έχουμε ενισχυμένη συνεργασία των υπηρεσιών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο με βελτίωση της συνέργειας, ε, με μεγιστοποίηση ε, όλων των δυνατοτήτων και ε, με ενισχυμένη συνεργασία με τρίτες χώρες προτεραιότητας προχωρούμε στα επιχειρησιακά μέτρα για την καταπολέμηση της διακίνησης μεταναστών. Ε, τα οποία συμπεράσματα ενέκρινε το Συμβούλιο το 2018, το Δεκέμβριο. Ενισχύονται ήδη κείμενα μέτρα στο πρόγραμμα δράσης κατά της διακίνησης μεταναστών 2015-2020 και έχουμε και νέες δραστηριότητες όπως κοινού συνδέσμους, ε, task force ε, με τη Europol. Ενισχύουμε επίσης την καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος με τη Europol ή ενισχύουμε τη δυνατότητα ε, να παρακολουθούμε και να διακόπτουμε τις ηλεκτρονικές διαδικτυακές επικοινωνίες των διακινητών. Στις 6 Δεκεμβρίου του 2018 εγκρίθηκε το, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ε, όπως ε, ίσως γνωρίζετε, ένα πρόγραμμα δράσης 10 σημείων. Ε, τέλος, ζητήσαμε να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία των τελωνίων στην εσωτερική ασφάλεια. Ε, η Βουλγαρική Προεδρία το Μάιο του 2018 έκανε μια θεματική σύσκεψη ε, για να ε, ενταχθούν τα τελωνία σε αυτή την προσπάθεια, να υπάρχει θεσμική συνεργασία, επιχειρησιακή συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς επίσης και διαλειτουργικότητα. Ε, για το σκοπό αυτό η Αυστριακή Προεδρία στη συνέχεια ε, ξεκίνησε κάποιες θεματικές ε, συζητήσεις μεταξύ των τελωνιακών αρχών. Η Κόζη καλωσόρισε την διάμεση έκθεση το Νοέμβριο του 2018 και ενθάρρυνε να συνεχιστούν οι εργασίες για τις προτεραιότητες αυτές του 18 μήνου. Οι συνέργειες λοιπόν και ευκαιρίες συντονισμού των δραστηριοτήτων και των πεπραγμένων στον κύκλο πολιτικής για το 2018 και διερευνήθηκαν και επίσης ε, ε, η ομάδα εργασίας η ένατη για τη συνεργασία με ε, τα τελωνία. Έχουμε πλέον και μια συνάντηση στις 26 Δεκεμβρίου 2018 αστυνομικών διευθυντών, επικεφαλής μάλλον των αστυνομικών υπηρεσιών και των τελωνίων για να υπάρξει πιο στενή συνεργασία μεταξύ αστυνομικών και τελωνιακών. Ε, τέταρτο θέμα, καταπολέμηση τρομοκρατίας. Προτεραιότητα παραμένει αυτή στην ατζέντα μας. Για το 2017, τον Νοέμβριο, ε, εγκρίναμε ε, ένα νέο τρόπο εκτίμησης της απειλής και του κινδύνου με στόχο να βελτιωθούν οι συστάσεις βάσει εκθέσεων της Europol και της ομάδα υψηλού επίπεδου για τη ριζοσπαστικοποίηση που θεσπίστηκε το 2017 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο να επιταχύνουμε τον τρόπο με τον οποίο ενημερωνόμαστε και ανταλλάσσουμε υποφορίες για τη ριζοσπαστικοποίηση των τρομοκρατών. Για να υπάρξει πολιτική και νομοθετικό πλαίσιο για να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατική απειλή σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις των τρομοκρατών και των επιστρεφόντων ε, Βουλγαρική Προεδρία ε, συνεργάστηκαν ομάδες εργασίας ΣΥΣΑ ΕΡΗΝ και ε, καταπολέμηση τρομοκρατίας για συγκεκριμένες συστάσεις που κατέληξαν σε συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ενίσχυση συνεργασίας στα ε, συστήματα SIS, Schengen Information System για ανθρώπους που συνδέονται με τρομοκρατικές εγκληματικές δραστηριότητες. Πέμπτη ενότητα. Το 2017 ε, εγκρίναμε τέσσερις συγκεκριμένες προτεραιότητες για την ε, πολέμηση ε, του dark web και του ηλεκτρονικού εγκλήματος μετά από μεγάλες κυβερνοεπιθέσεις. Βελτιώνουμε τη δυνατότητα διερεύνησης τώρα του ε, οργανωμένου εγκλήματος στο διαδίκτυο. Καθόλου το 18 μήνο επίσης. Έκτη ε, ενότητα και τελευταία σχέση εσωτερικής εξωτερικής ασφάλειας. Αυτό εξακολουθεί να μας ε, απασχολεί πάρα πολύ ε, κάθε εξάμεινο έχουμε κοινέ συνεδριάσεις με την άλλη αρμόδια επιτροπή και ένα πιλωτικό πρόγραμμα, ε, μια μονάδα για ενημέρωση σχετικά με το έγκλημα στην επιχείρηση Σοφία ε, βοήθησε πάρα πολύ για τη βελτίωση της επιχειρησιακής συνεργασίας της ΕΠΑ, της εξωτερικής πολιτικής και της εσωτερικής πολιτικής και πολιτικής δικαιοσύνης. Ξέρουμε ποιο ρόλο έχει ο καθένας και ποια ευθύνη. Παρακολουθούμε ε, και τι γίνεται στο πολιτικό σκέλος της ΕΠΑ, της Εξωτερικής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας, για να συνδέσουμε καλύτερα την εσωτερική με την εξωτερική ασφάλεια. Να διευρυνθεί η, το πεδίο εφαρμογής των πολιτικών μη στρατιωτικών αποστολών στις 19 Νοεμβρίου του 2018 το ενέκρινε αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είναι σημαντικό να υποστηρίζουν αυτή την προτεραιότητα και την πρωτοβουλία τα κράτη-μέλη με εθνικά σχέδια ε, αυτό τονίστηκε. Κατά τη διάρκεια τη Ιστονικής Προεδρία, η ΚΟΖΗ προετοίμασε τις συμπεράσματα του Συμβουλίου για την εξωτερική ε, συνεργασία και συνεργασία εσωτερική ασφάλειας με την Ουκρανία που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 2017. Έδειξαν οι συζητήσεις ότι χρειάζεται να υποστηριχθούν οι διοκτικέ αρχέ, ιδιαίτερα μέσω τη ΕΠΑ στην Ουκρανία. Τον Ιούνιο του 2018 ενημερώθηκε η ΚΟΖΗ από τους επικεφαλείς της αποστολής στην Ουκρανία. και χρειάζονται ε, πέντε τομείς ε, υποστήριξης για τη δημόσια τάξη, για τις ε, έρευνες που γίνονται στα κλίματα. Η συνεργασία με τα Βαλκάνια επίσης κυριάρχησε το τελευταίο 18 μήνο. Είναι πολλές οι περιφερειακές δραστηριότητες. Η Επιτροπή μας κόζει τόνισε τη σημασία να ενταθούν οι προσπάθειες στην περιοχή ε, όπου θα μπορούσε να αξιοποιηθεί πλήρω ο ρόλο των οργανισμών δικαιοσύνη και εσωτερικών. Δηλαδή να ενισχυθούν τα δίκτυα των επαγγελματιών του κλάδου, των εργαζομένων σε αυτούς, για να μειώνονται οι περιφερειακές εντάσεις, οικοδομείται εμπιστοσύνη και συνεργασία αυτό το τονίζεται και ο κύκλος πολιτικής και μπορεί να αποτελέσει μια γερή πλατφόρμα για τη συνεργασία μας, την ενισχυμένη συνεργασία στα Δυτικά Βαλκάνια. Αξιότιμοι βουλευτές, σας ευχαριστώ και πάλι που μου δώσατε την ευκαιρία να απευθυνθώ στην Επιτροπή σας για τα θέματα αυτά και με χαρά να απαντήσω σε ερωτήσεις που τυχόν θα είχατε. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτή. Ε, μου επιτρέπετε να ξεκινήσω με κάποια σχόλια εγώ και κάποιες ερωτήσεις. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω που ήρθατε εδώ και μας δώσατε κάποια στοιχεία για το έργο σας. Και η πρώτη μου ερώτηση είναι πολύ γενικής φύσεως. Με βάση την εμπειρία σας σύντοχρον θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε ιδιαίτερα επειδή συζητούμε για τις τρομοκρατικές ε, επιθέσεις στην Ευρώπη και την ε, αυριανή μέρα, υπάρχει συζήτηση για το πώς μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών αλλά και ευρωπαϊκών οργανισμών. Υπάρχει καλύτερη συνεργασία, υπάρχει καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών, κάποια σχετική συζήτηση. Αυτή είναι μια γενική ερώτηση, όπως είπα. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στο διαδικτυακό έγκλημα που αναφέρατε είναι μια άλλη έκφραση για το κυβερνό έγκλημα έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Μπορούμε να έχουμε κάποια παραδείγματα, γιατί με του ορισμού κάποιε φορέ δημιουργείται σύγχυση και δεν καταλαβαίνουμε περί τίνο πρόκειται. Και μια τελευταία δική μου παρατήρηση. Μιλήσατε, αν δεν απατώμε, για έξι προτεραιότητε που επεξεργάζεστε και δίνετε μια συνέχεια σε όλο το έργο που έχετε κάνει. Έχετε εραρχήσει αυτά τα σημεία, τα έξι χρειάζονται για κάποια περισσότερες δράσεις ή είναι όλα στο ίδιο επίπεδο. Παρόντω αυτά, θα μπορούσα να προσθέσω και άλλε ερωτήσει. Απαντήστε όμω πρώτα σε αυτέ τι τρει ερωτήσει. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Ε, απάντηση. Σα ευχαριστώ πολύ. Σε ό,τι αφορά την τρομοκρατία, ίσως το σημαντικότερο είναι το θέμα της διαλειτουργικότητας, Οι δέσμοι μέτρων για τη διαλειτουργικότητα και η βάσεις ε, δεδομένων όπως πηγαινά, αρέτειας, που θα αλλάξουν τα δεδομένα στις ε, ε, αρχές επιβολής του νόμου. Βλέπουμε ότι το είδαμε και στις πρόσφατες επιθέσεις, ότι υπάρχουν κάποιοι που ταξιδεύουν και παίρνουν από πολλές χώρες. Σίγουρα λοιπόν πρέπει να συναντώμεθα και να συζητούμε. Αυτό είναι όλο και πιο επίκαιρο, όλο και πιο σημαντικό. Εξού και όλες οι προεδρίες συνεργάστηκαν για την εκπόνηση αυτή τη έκθεση επί Ρουμανική Προεδρία. Επίση, να σα πω ότι όλε οι προτεραιότητε αποσκοπούν στην ε, δημιουργία γεφυρών μεταξύ των διαφόρων εμπλεκομένων φορέων. Μιλάμε δηλαδή για κρατημέλη, για οργανισμού ε, δικαιοσύνη εσωτερικών θεμάτων, αλλά και πολλού ε, επαγγελματίε των διαφόρων κλάδων στην ομάδα εργασία Χάρη για την επιβολή τη νομοθεσία. Και υπάρχουν διάφορα project που εντοπίζουν τρόπου, μεθόδου, διαδικασίε για την κατανόηση τρομοκρατία, για την εξέβρεση τρόπων αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού. Συζητούμε για διάφορα project μεταξύ αυτών και τα χρηματοδοτούμενα από την Ένωση. Και γενικώ πρέπει να σα πω ότι αυτό είναι μια, φρέ... είναι μια νέα ανάσα για του οργανισμού αυτού επιβολής του νόμου. Από την Γερμανική Προεδρία, μια από τις πρωτοβουλίες μας λέγεται πρόσβαση στην πληροφορία. Γιατί για μας είναι πολύ σημαντική η πληροφόρηση, άρα θέλουμε να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα ανταλλαγή πληροφοριών για την εισίδες γνώσης και για την καταπολέμηση της ε, τρομοκρατίας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ενίοτε όμως πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη προβολή και να μην ξεκινάμε από το μηδέν κάθε φορά για να επανεφεύρουμε τον τροχό. Καλό θα ήταν να ξέρουμε πού οι προηγούμενοι σταμάτησαν και συνεχίσουμε εμείς και να βελτιώσουμε τις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναλυφθεί. Γι' αυτό λοιπόν δημιουργήσαμε αυτή την πλατφόρμα που ε, υπάρχει μια συγκέντρωση ε, δεξιοτήτων, εμπειριών και η εμπειρία μιας χώρας μπορεί να βοηθήσει σε μια άλλη περίπτωση σε ένα κράτος μέλος που ένας πάρα πολύ έτσι, δραστήριος και ενθουσιώδης πάλι μπορεί να αντλήσει χρήσιμες πληροφορίες. Γιατί λοιπόν να ξεκινάμε πάντα από την αρχή και το, εννοώ, το λέω και για τους χαράκτες πολιτικής και για τους ε, αστυνομικούς διευθυντές. Καλό είναι να υπάρχει συνεργασία για να ξέρουμε πού πάμε και να μην πηγαίνει ο καθένας από μόνος του. Αυτές είναι οι τελευταίες τάσεις και οι απαντήσεις. Δίκτυα, κράτη-μέλη και φορείς Δικαιοσύνη και εσωτερικών θεμάτων συνεργάζονται σε ό,τι αφορά το διαδικτυακό έγκλημα και σε σχέση με το έγκλημα στο κυβέρνοχώρο. Αυτά τα συζητούν τα κρατημέλη και οι διάφορες υπηρεσίες. Όταν αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα του έγκληματος στον κυβέρνοχώρο, θεώρησαμε ότι ίσως να μην αφορά τους πάντες. Είναι συγκεντρωμένες, στοχευμένες επιθέσεις σε μια επιχείρηση ή σε κάποιο ιδιώτη. Και είπαμε να συγκροτήσουμε ομάδε ολιγομελεί μεν, που όμω ε, θα είναι πολύ καλέ σε αυτό που κάνουν, δηλαδή να κατανοήσουν το φαινόμενο του εγκλήματος στον χώρο. Όμω, τι είδαμε την τελευταία δεκαετία. Όλα κινούνται προ το διαδίκτυο. Για παράδειγμα, θέλω να ε, το αυτοκίνητό μου. Πριν 10 χρόνια για να το κάνω αυτό θα έβαζα μια αγγελία σε μια εφημερίδα, ενώ τώρα θα τη βάλω στο διαδίκτυο. Το ίδιο αν θέλει κάποιο να πουλήσει το πλυντήριό του να αγοράσει κτλ. κτλ. Αν είμαι λοιπόν θύμα απάτη όταν προσπαθώ να πουλήσω μέσω, του, μέσω, ε, μέσα από το διαδίκτυο αυτοκινητό μου. Αυτό δεν είναι κυβερνό έγκλημα. Τι κάναμε λοιπόν στο παρελθόν και κάνουμε ακόμη και τώρα ενίοτε. Χρησιμοποιούμε αυτού του επαείοντε για την καταπολέμηση του κυβερνοκλήματο και για να ερευνήσουν εγκλήματα που συμβαίνουν μέσα στο διαδίκτυο. Και επειδή όλα ε, μπαίνουν στο διαδίκτυο, Πολλέ επιχειρήσεις μπαίνουν στο διαδίκτυο και υπάρχουν και νομοθετικέ πτυχές, οι πτυχές που άπτονται τη ανοιχτή διακυβέρνηση, της διαφάνειας κτλ. Η τάση αυτή είναι, πρέπει να την παρακολουθούμε και πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να δημιουργήσουμε περισσότερες ομάδες για την αντιμετώπιση αυτού του είδους ε, εγκλήματος η αφρόκρεμα της έρευνας θα είναι σίγουρα ο κυβερνοχώρος και τα εγκλήματα εκεί. Όμως πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τα εγκλήματα τα κοινού ποινικού δικαίου, εγκλήματα στο διαδίκτυο και τις σχετικές αξιόπινες πράξεις. Και ο Ντεμπόλ έκανε μια παρουσίαση προηγουμένως και είπε πολλά. Και συνεργαζόμαστε. Η Europol βοηθάει ιδιαίτερα να καταλάβουμε τη διαδικότητα αυτή και τη σχέση διαδικτυακού και κυβερνογκλήματος. Και υπάρχει και αυτή η πλατφόρμα, όπως είπα, ανταλλαγής πληροφοριών που θα φιλοξενηθεί από τη Europol. Αυτό θα είναι και το βασικό μας εργαστήριο. Σε ό,τι αφορά τις έξι προτεραιότητες, έπρεπε να τις καταγράψουμε η ασφάλεια και καταπολέμηση του κλίματος. Είναι πολύπλοκοι στόχοι και αλληλένδετοι. Ευχαριστώ αυτά. Thank you very Ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις ε, επιπλέον ερωτήσεις, Ε, ερώτησα, ερώτησα τι ιεράρχηση θα μπορούσε να υπάρχει σε αυτές τις έξι προτεραιότητες, γιατί το πρώτο που αναφέρατε είναι η καταπολέμηση των λαθρομεταναστών, δηλαδή της εμπορίας και της λαθρομετανάστευσης και μετά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Εγώ σκέφτηκα ότι ίσω η απειλή τη τρομοκρατία να μην είναι πια τόσο σημαντική. Ε, όμως σωστά και εσείς είπατε ότι όλα είναι αλληλένδετα μεταξύ τους. Δεν βλέπω να ζητά άλλο κανεί να θέσει ερωτήσει. Καταλαβαίνουμε λοιπόν όλοι ότι η δουλειά τη ΚΟΖ είναι πολύ σημαντική, η συνεργασία είναι πολύ σημαντική. Καταλαβαίνω ότι αυτή η σχετικά νέα πλατφόρμα για την ανταλλαγή των πληροφοριών είναι πολύ σημαντική, αλλά πραγματικά για ανταλλαγή γνώσεων, ε, στοιχείων για τους ανθρώπους που μας ενδιαφέρουν. Είναι κάτι του πολύ θετικό. Λίγο με ανασυχεί η οπτική αναγνώριση, η αναγνώριση βάσει του προσώπου. Δεν είναι κάτι που το είχαμε αποφασίσει εδώ, αλλά μπορούμε να το συζητήσουμε και στο μέλλον. Διότι στον ψηφιακό μας κόσμο πρέπει να μπορούμε να αξιοποιήσουμε ό,τι είναι διαθέσιμο. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ και καλή τύχη ε, για την δουλειά σας στο μέλλον. So, Λοιπόν, το επόμενο θέμα κανονικά στην ημερήσια διάταξή μας είναι η ηλεκτρονική ψηφοφορία, η οποία έχει προβλεφθεί δυστυχώς για τις 5 και 4. Τι να κάνουμε τώρα, δυστυχώς μάλλον θα πρέπει να διακόψουμε και ελπίζω να έχουν έρθει όλοι οι συνάδελφοι για να ψηφίσουμε στις 5 και 4 για αυτό το θέμα της συμφωνίας με τη Δανία για την Eurojust. Έχετε την ευκαιρία να κάνετε ένα διάλειμμα τώρα, να πάρετε κανένα καφέ, να βγείτε έξω να δείτε λίγο ήλιο, γιατί από εδώ δεν βλέπουμε το φως της μέρας. Θα τα πούμε στις 5 και 4.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

Yeah. να κάνεις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

Uh, so, colleagues, colleagues, we just begin the uh, meeting. Um, Συνάδελφοι, αρχίζουμε τη συνεδρίασή μας που έχει μία ψηφοφορία και μετά θα πάμε στην κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Έτσι δεν είναι. Ωραία. Ένα θέμα έχουμε να ψηφίσουμε. Θα πρέπει να σας ε, αναφέρω τα αποτελέσματα των συντονιστών Αποφάσισα να αλλάξει εισηγητής για το θέμα ε, του Brexit. Ο κύριος Τανίσεφ ε, το αναλαμβάνει αυτό και το υλικό τριμερής διάλογος θα λάβει χώρα αύριο για τις θεωρήσεις μετά το Brexit. Έχουμε το σημείο 5α, ψηφοφορία για τη Eurojust 5α, το ζήτησε η πολιτική ομάδα των φιλελευθέρων. Ε, βάσει του άρθρου 205. Πολύ σύντομα πριν ψηφίσουμε. Εδώ περιμένουμε την, ε, το σχέδιο συμφωνίας που θα υποβληθεί για την επόμενη ε, θητεία. Πριν όμως ψηφίσουμε για την αναβολή, να θυμίσω, για να είμαστε ξεκάθαροι, ότι αν είστε υπέρ της σύστασης των συντονιστών, για αναβολή θα ψηφίσετε Plus. Εάν είστε υπέρ τη σύσταση για την αναβολή Plus, εάν είστε κατά τη σύσταση των συντονιστών, θα βάλετε μείον. Ή βεβαίω μπορείτε και να απόσχετε. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονική. Εψήφισαν άπαντε. Άρχεται. Εάν είστε υπέρ, συν, εάν είστε κατά, μείον. Άρχεται η ψηφοφορία. Has everyone voted? The vote is closed. Πέρας. Εψήφισαν άπαντες. Η απόφαση των συντονιστών ε, με 16 ψήφους προς 4 απορρίπτεται και καμία αποχή. Και τώρα που απορρίφθηκε θα ακολουθήσουμε την ταχεία διαδικασία, μόνο αγγλικά. Προεδρεύω, παρακαλώ να μπει υποσημείωση, παρουσίαση του σχεδίου συμφωνίας στις 8 Απριλίου, ψηφοφορία στην ΛΥΜΠΕ. Αρκεί να είμαι και εγώ εδώ που θα είμαι στις 8 Απριλίου. Και μετά θα περάσει και στην Ολομέλεια τη δεύτερη του, του Απριλίου. Εδώ θα είμαι όμως ακόμα καλό αυτό, οπότε καταλαβαίνω ότι οι περισσότερες πολιτικές ομάδες έχουν πει ότι θα έπρεπε να είμαι ο ε, εισηγητής ως, ε, λόγω της θεσμικής μου δυνατότητας. Συμφωνείτε? Κάντε κάποιο νεύμα της ε, θεσμικής μου ιδιότητας. Εδώ λοιπόν στις 3 θα παρουσιαστεί το σχέδιο στην Επιτροπή ΛΥΜΠΑ τέλος αυτού του μέρους της συνεδρίασης και τώρα πάμε στο 1G3, στο ASP, ε, κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Θα σας δω εκεί.